Witam koleżanki i kolegów. Otwieram sesję przerwaną w dniu 23 czerwca. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ξεκινήσουμε τη, ξεκινούμε τη συνεδρίαση συνεχίζοντας μετά τη διακοπή τη 24 η Ιουνίου του 2010 τα πρακτικά των κειμένων ε, που ε,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 σε θανατική ποινή και ενώ αυτά τα παιδιά τώρα έχουν πλέον ελικιωθεί, βρίσκονται στην ε, φυλακή περιμένοντας την εκτέλεση της θανατικής τους ε, ποινής. Στις 13 Ιουλίου επίσης ε, μνημονεύσαμε την επέτειο του θανάτου του Γιάννη Κάρσκι ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος συνέταξε έκθεση προς τους συμμάχους για το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 ε, βουλευτών και των νέων θέσεων που αναλαμβάνουν σε επιτροπέ και αντιπροσωπείε. Εάν δεν υπάρχουν και από την ομάδα των φιλελευθέρων επίση, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θεωρούμε ότι έχει εγκριθεί αυτό ο κατάλογο των ορισμών για τον προπολογισμό. για την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 Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι για μας είναι η έκθεση όριμη προς ψήφιση. Όπως λέμε, τα φρούτα πρέπει να τα κόβουμε όταν είναι όριμα, όχι όταν είναι άγουρα, ούτε, ούτε όταν είναι σάπια. Για μας είναι όριμο λοιπόν και πρέπει να ψηφιστεί. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε κυρίε και κύριοι. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για αναβολή της έκθεσης. Καλό. Παρακαλώ σηκώστε τα χέρια. Ευχαριστώ. Κατά. Θα κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Η πρόταση εγκρίνεται. Η έκθεση «Καλό» αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Για την Τρίτη και την Τετάρτη δεν υπάρχει καμία πρόταση τροποποίησης. Σε ό,τι αφορά την Πέμπτη, οι Ευρωπαίοι μεταρρυθμιστές προτείνουν να συζητηθούν οι περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου την Πέμπτη το απόγευμα με τον εξής τρόπο. Πρώτον, υπάρχει μία πρόταση για τη Ζιμπάμπουε, τη Βενεζουέλα και τη Βόρεια Κορέα. Προτείνεται να, να αντιστραφεί η σειρά. ο σκάλα να έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να το αίτημά μα να μην είναι δύσκολο και ποιημάχο απλώ να προσαρμοστεί κάπω σήμερα στη διάταξη την Πέμπτη απόγευμα στη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε το Ζιμπάμπου να συντηθεί πρώτα, μετά η Βενεζουέλα, μετά η Βόρεια Κορέα. Δεν κάνουμε καμία προσπάθεια να δώσουμε οποιαδήποτε σημασία ιδιαίτερη σε κανένα αυτά τα θέματα. Απλώ βολεύει, εάν εξεταστεί πρώτα το θέμα τη Ζιμπάμπου, βολεύει κάποια μέλη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ψηφίσουμε λοιπόν αυτή την πρόταση. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει υπέρ της προτάσεως. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως υπεγράμμισε και ο συνάδελφος, εδώ δεν πρόκειται περί εισαγωγής ή αφαιρέσεως θεμάτων από την ημερήσια διάταξη, αλλά απλώς να αντιστραφεί κάπως η θέση να αλλάξει θέση των διαφορών θεμάτων που θα πρέπει να συζητηθούν. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η πρόταση μπορεί εύκολα να γίνει αποδεκτή. Πρόεδρος, υπάρχει κάποιος που επιθυμεί να πάρει το λόγο και να μιλήσει κατά της προτάσεως αυτής. Έχετε το λόγο. Κύριε Σούλτς, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου μια ερώτηση προς τον αγαπητό συνάδελφο Κέλλεναν. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί εξυπηρετεί του συναδέλφου σας να συζητηθεί πρώτο το θέμα της Ζιμπάμπουε και ποιους εκ των συναδέλφων σας εξυπηρετεί αυτό. Είναι σημαντικό κριτήριο αποφάσεως για μας. Γιατί λοιπόν, θέλετε να μας πείτε. Ποιος είναι ο ιδιαίτερος λόγος που θέλετε να έρθει μπροστά στο πρόγραμμα Ζιμπάμπουε, γιατί σας διευκολύνει να τη συζητήσουμε πρώτη. Πρόεδρος. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Σούλτς με βάζει πολύ δύσκολη θέση. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Απλώς διαβιβάζω το αίτημα συναδέλφου του κυρίου Βανόρντεν, ο οποίος καθυστέρησε και κάποιος μου ζήτησε αν έχω την καλοσύνη να το θέσω το θέμα εκ των προτέρων. Γι' αυτό. Όπως πάντα η καλύτερη πολιτική είναι η ειλικρίνεια με τον κύριο Σούλτ. Πρόεδρος. Εν τη αυτή περιπτώσει ας ψηφίσουμε. Ποιο είναι υπέρ αυτής της προτάσεω, Σας σηκώστε το χέρι παρακαλώ. Σας ευχαριστώ.